και ε, η πρωτοβουλία για το κέρας της Αφρικής με δηλώσεις Συμβουλίου και Επιτροπής. Δίνω μέσω στο λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου στον ε, Υπουργό τον κύριο Ντελα Βέντοβα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Με μεγάλη χαρά απαντώ σε αίτημα για δήλωση του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής σε θέματα μεταναστευτικών οδών, όπως αποκαλείται διαδικασία της Χαρτούμ και συγκεκριμένα σε σχέση με τα πορίσματα της Υπουργικής Διάσκεψης που έγινε στη Ρώμη στις 28 Νοεμβρίου του 2014. Θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου ικανοποίηση, αλλά και την ικανοποίηση της Προεδρίας για την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στην διάσκεψη αυτή που ήταν θεμελιώδης για να είναι αυτή επιτυχής. Συμφωνούμε όλοι για το γεγονό ότι η συνεργασία με τι χώρε προέλευση και διέλευση των μεταναστών σε ένα πνεύμα διαλόγου εταιρική σχέση και κοινή ευθύνη είναι σημαντική ουσιαστική για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η διαδικασία του χαρτόμο, που θεσπίζεται, θεσπίστηκε στη διάσκεψη της Ρώμης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ένα πλαίσιο εντό του οποίου μπορούμε να συζητήσουμε την μετανάστευση και τα σχετικά θέματα με διάφορου σημαντικού εταίρου τη Ανατολική Αφρική. Μετά από μια σειρά άκαρπων απόπειρων, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη καταφέρουν να ξεκινήσουν έτσι μια διαδικασία σε θέματα μετανάστευση. Αυτό σημαίνει πω θα είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε έναν τακτικό διάλογο με τι χώρε του κέρατο τη Αφρική και τη Ανατολική Αφρική περιοχέ Προέλευση, διέλευση και σημαντικών μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημαντική αύξηση των αφήξεων μεταναστών από την ε, περιοχή αυτή και από την κεντρική ε, μέσω της Μεσογείου ε, προκύπτει λόγω της κατάστασης της περιοχής και λόγω της ύπαρξης ε, διαδρομών που χρησιμοποιούνται από τους μετανάστες. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην καταπολέμηση της δουλεμπορίας. Η δήλωση που υιοθετήθηκε από τη διεπουργική αυτή διάσκεψη ε, υποδεικνύει διάφορα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν και όλοι γνωρίζουμε πως πρέπει επιγόντως να ληφθούν μέτρα για να μπορέσουμε να διώξουμε ε, τους ε, δουλέμπορους και να διαλύσουμε τα δίκτυά τους. Ο στόχο, όπω υπογραμμίζει σαφώ η δήλωση, είναι να φτιάξουμε ένα διάλογο που θα συμπεριλαμβάνει όλου του τομεί που καλύπτει η σφαιρική προσέγγιση σε θέματα μετανάστευση και κινητικότητα. Νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα, παράνομη μετανάστευση, μετανάστευση και ανάπτυξη, διεθνή προστασία. ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσω ότι η δήλωση αναγνωρίζει την προώθηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ω θέματα τα οποία διέπουν τη συνεργασία μας. Επίσης αναγνωρίζει ρητά την ανάγκη να γίνουν σεβαστά και να ενημερωθούν, να εξυγχρονιστούν οι αρχές της διεθνούς προστασίας με σαφή αναφορά στη Σύμβαση της Γενέβης του 1951. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, έχουμε ορίσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασία για τη διαδικασία του Χαρτούμ και νομίζω πω πρόκειται για μια καλή αρχή. Ξεκινώντα με αυτή τη βάση, είναι η στιγμή να περάσουμε σε μια πιο δραστήρια φάση. Καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη τη να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση αυτή τη νέα διαδικασία. Η στήριξη αυτή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία τη Χαρτούμ θα είναι θεμελιώδη για την επιτυχία και την αίσια της έκβαση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος, κύριε Υπουργέ. Ακολουθεί η Κομισιόν. Κύριε Αβραμόπουλος, σας δίνω το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μέλη του Κοινοβουλίου. με έχετε κάνει να ταξιδέψω από την, τις Ηνωμένες στη Γεωργία και από την Γεωργία στο κέρας της Αφρικής. Νομίζω ότι αυτές οι μετακινήσεις όμως έχουν μεγάλη σημασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δει στις συζητήσεις που έχει διαξαγάγει το πόσο σημαντικό είναι να σώσουμε τις ζωές αυτών που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Μέσα και σε αυτή την αίθουσα έχω ακούσει επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να δώσουν πρακτικές απαντήσεις στην πολιτική πραγματικότητα της λαθεμπορίας μεταναστών και της εμπορίας ανθρωπίνων όντων από το κέρας της Αφρικής. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο διαλόγου και ένα πλαίσιο εφαρμογής λύσεων μαζί με τις χώρες της περιοχής. Αυτό είναι η πρωτοβουλία για τη μετανάστευση Ευρωπαϊκής Ένωσης του κέρατος και του κέρατος Αφρικής μια πολιτική ε, πρωτοβουλία διαλόγου με τις χώρες αυτές της, ε, του κέρατος Αφρικής και, τους, και τις χώρες διέλευσης προς τη Μεσόγειο. Οι χώρες λοιπόν <clears throat> προέλευσης, διέλευσης και προορισμού πρέπει να έρθουν από κοινού για να συζητήσουν τα θέματα αυτά. Οι χώρες αυτές τις, ε, που εμπλέκονται είναι το Τζιμπουτί, η Αίγυπτος, η Ερυθρέα, η Αιθιοπία, η Κένια, η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και το Σουδάν, αλλά και η Λιβύη και η, Λιβύη και η Πέραν λοιπόν των απλών πολιτικών δηλώσεων, πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές θα πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα επιβολής του νόμου στις αφρικανικές χώρες ώστε να καταπολεμηθούν οι λαθρέμποροι και οι δουλέμποροι με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν ε, σημαίνουν μόνο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες τόσο για τις χώρες προέλευσης όσο και για τις χώρες προορισμού. Γι' αυτό ακριβώς και πιστεύω ότι η συνεργασία μας με τις χώρες εταίρου σε αυτή τη διαδικασία δεν θα πρέπει να σταματά στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Θα πρέπει να φτιάξουμε, να, να θέσουμε ψηλές φιλοδοξίες και να εξετάσουμε από κοινού ποιε είναι οι ρίζες των μεταναστευτικών φαινομένων. Εσείς, οι αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Έχετε οι ίδιοι ζητήσει την εξασφάλιση επατολισματικής συνεργασία με τρίτε χώρε προέλευση, αλλά και διέλευση για τον σκοπό αυτό. Το κέρας της Αφρικής και η σχετική πρωτοβουλία είναι μια από τις απαντήσεις, που θέλουμε να δώσουμε σε αυτές τις εκκλήσεις σας. Σύμφωνα με τη δήλωση για την ε, μετανάστευση και την κινητικότητα που υιοθετήθηκε από τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων στην τέταρτη σκέψη κορυφή Ένωσης Αφρικής, λένε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε την ανάπτυξη αλλά και τις ευκαιρίες νόμιμης μετανάστευσης καθώς και να μεριμνήσουμε για αποτελεσματική διεθνή προστασία των όσων τη χρειάζονται. Η πρωτοβουλία μετανάστευσης της Αφρικής μπορεί να μας βοηθήσει ε, να να συνειδητοποιήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να δούμε τις υπήρους μας σε ένα πνεύμα κοινή ευθύνη. Ξέρω ότι πολλοί στο σώμα έχουν απορίες για το πώς τα ανθρώπινα δικαιώματα να περιλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα σε χώρες όπου οι δημοκρατικές αξίες δεν γίνονται σεβαστές. Μπορώ να σα να σας διαβεβαιώσω πως το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει προτεραιότητα στην μεταναστευτική μα πολιτική και την εξωτερική της διάσταση και αυτό αντικατοπτρίζεται απόλυτα σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου. Από αυτή τη βάση μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτή τη διαδικασία και να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει και θα προσαρμόζεται διαρκώς στους πολιτικούς μας στόχους. Στόχους κοινούς, απόλυτα αποδεκτούς και εθελοντικούς. Προσβλέπω σε μια ομαλή κίνηση πρακτικών δράσεων και σχεδίων ώστε αυτό ο διάλογος να τεθεί σε πράξη, να, να μετατραπεί σε πράξη και να επιτύχει απτά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στα δύο κεντρικά θεζητήματα που είναι η <coughs> δημιουργία στρατηγικής για την εθελοντική επιστροφή και ενσωμάτωση των μεταναστών. Με χαρά ανακοινώνω ότι για αυτό το στόχο αρχική χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ έχει ήδη εντοπιστεί από το ε, όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή βοήθεια επίση επίσης να αναπτυχθούν ε, ε, οργανωμένες δράσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα το λαθρεμπόριο και την δουλεμπορία. <coughs> Ε, έχουμε βάλει στην άκρη 750.000 ευρώ από το Διεθνές Ταμείο Ασφάλειας για να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δράσεις. Οι κόρες, τα προγράμματα αυτά τώρα είναι η στην Κομισιόν και η εφαρμογή του θα ξεκινήσει του χρόνου. Θα ενθαρρύνουμε τους εταίρου μα από την Αφρικανική Ήπειρο να εξετάσουν αυτές τις προτάσει και να βοηθήσουν στην εφαρμογή τους. Τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να παίξουν ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή αυτή τη πρωτοβουλίας σε σχέση με τους δύο αυτού χώρους που προανέφερα. Πρέπει να υπάρξουν ε, ενίσχυση των σχέσεων και του διαλόγου και να προωθήσουν λύσεις οι οποίες θα έχουν με βιώσιμο και μόνιμο χαρακτήρα. Είναι λοιπόν στα χέρια μας το να βελτιώσουμε την κατάσταση σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Νομίζω ότι η δημιουργία ενός βιώσιμου διαλόγου και η επίτευξή του με συγκεκριμένες ενέργειες επιτόπου θα είναι η λύση. Πρέπει να δράσουμε τώρα <clears throat> και πρέπει να δράσουμε από κοινού. Μόνο με το να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα δάξουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Η Κομισιόν βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πολιτική υποστήριξη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημαντική σας τοποθέτηση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών του ομάδων. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για 1,5 λεπτό η κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω τη διαδικασία του Χαρτούμ που εκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες. Η διαδικασία αυτή έχει στόχο την καταπολέμηση του δουλεμπορίου, της διακίνησης μεταναστών από το κέρας της Αφρικής προς την Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή ενθάρρυνει τις χώρες να καθίσουν από κοινού στο ίδιο τραπέζι και να ξαναρχίσουν το διάλογο. Έχουμε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε πει επανειλημμένα και το ξαναλέω σήμερα. Ο μόνος δρόμος για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική περνάει <coughs> μέσα από σφαιρικές καθολικές λύσεις που ε, εξετάζουν όλες τις πτυχές και μία από τις πιο σημαντικές πτυχές είναι να εξασφαλίσουμε την πλήρη μας συνεργασία με τρίτες χώρες της Αφρικής, ιδιαίτερα με τις χώρες προέλευσης αλλά και τις χώρες διέλευσης. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις χώρες για την καταπολέμηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας στην οποία πέφτουν θύματα ε, οι πιο ευάλωτοι. Θα πρέπει να δούμε και τις ρίζες και τις αιτίες του κακού. Τι οθεί τους ανθρώπους να φεύγουν από την πατρίδα τους. Ε, όλα αυτά λοιπόν είναι ε, πολύ σημαντικά και μια ευρεία διαδικασία για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα θύματα αυτής της παρανομίας, αυτού του εμπορίου ανθρώπων. Πρέπει να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ζωές των μεταναστών που πέφτουν θύματα του τράφικινγκ. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και η απαραίτητη χρηματοδότηση για να αποδώσει η διαδικασία. Δεν μπορούμε απλούστατα να τη βάλουμε στο αρχείο ή σε ένα σιρτάρι τη διαδικασία. Πρέπει να υλοποιηθεί και να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και... Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Από την κυρία Βερζιά. Τη δέχεστε την ε, ερώτηση αυτή, κυρία Ματσόλα. Κυρία Βερζιά. Κυρία Μέτσολα, θα ήθελα να ξέρω αν γνωρίζετε την κατάσταση στις χώρες του κέρατος της Αφρικής και αν ξέρετε ποιος είναι ο ρόλος αυτών των χωρών στη λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων στην περιοχή αυτή. Κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ κυρία Βέζια. <clears throat> ναι, τη γνωρίζω την κατάσταση στις χώρες αυτές και έρχομαι και από μια χώρα η οποία υφίσταται ισχυρά αναστευτικά ρεύματα από τις χώρες αυτές και οι οποίοι ζητούν τη βοήθειά μας και έρχονται φυσικά από τις χώρες του κέρατος της Αφρικής. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα αγωνιστούμε εναντίον της ε, λαθρεμπορίας ανθρωπίνων όντων και να προστατεύσουν τα πιο τροτά από αυτά τα άτομα. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος <clears throat> για τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Η Μπίργκετ Ζίπελ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το να καταλάβουμε τους λόγους της μετανάστευσης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό η διαδικασία του Χαρτούμ είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ανοιχτά ερωτήματα. Το να αντιμετωπίσουμε τους ε, παράνομους διακίνητες πρέπει να είναι η μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και η προστασία των ανθρώπων που φεύγουν από τον πόλεμο και την πολιτική καταδίωξη. Η <clears throat> προτεραιότητα αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί με τη δημιουργία κέντρων κράτησης. Ορισμένοι λένε ότι είναι κέντρα φυλάκισης. Αλλά ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Θεμάτων λέει κέντρα υποδοχής. Το θέμα είναι πόσο καλό δεκτή νιώθουν αυτοί οι μετανάστες σε αυτά τα κέντρα. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι σημαίνει πρόσβαση στην ε, δυνατότητα να υποβάλουν μια αίτηση ασύλου και ποια είναι τα κριτήρια τα οποία ισχύουν για τις αιτήσει αυτές ασύλου. Θα είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν οι χώρες αυτές όπου βρίσκονται ή αυτά που θα καθορίσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μια πλήρη αίτηση ασύλου ή θα είναι απλώς ένα φράγμα για να αποθεί τα άτομα αυτά από την Ευρώπη. <clears throat> Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί η αρχή της ατομικής δυνατότητας υποβολής ασύλου. Η διαδικασία λοιπόν του Χαρτούμ θα πρέπει να τεθεί κάτω από μια πολύ κριτική αντιμετώπιση από τη δική μας πλευρά. <clears throat> θα πρέπει όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής να συμμετάσχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Γίνεται κάτι τέτοιο και επίσης είναι ποιος είναι ο ρόλος της Κομισιόν στην διαδικασία του θα υπάρξει <clears throat> μια χρηματοδότηση αυτής της διαδικασία σχετικά και πώς θα συμμετάσχει και πώς θα πληροφορείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα. Ελπίζω ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα μπορέσουν να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις σήμερα. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ η κυρία ε, Βίξτρομ από τη Φιλελεύθερη Ομάδα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Βίξτρομ, στα, στα πολωνικά. Είναι πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι θέλουν να πάνε στην Ευρώπη και να δημιουργήσουν μια νέα ζωή για αυτούς. Αλλά αντιμετωπίζουν, <clears throat> αντιμετωπίζουν πέρα από τις διώξεις της χώρες τους, αντιμετωπίζουν και το στίγμα του παράνομου. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν όμως καμία άλλη επιλογή παρά να βάλουν τον εαυτό τους στα χέρια των διακινητών, οι οποίοι τους βάζουν σε κάποιο σκάφος <clears throat> όπου θα κινδυνεύσουν τη ζωή τους για να φτάσουν στην Ευρώπη. 3.419 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο φέτος. Μόνο στη Μεσόγειο. Βάσει τι έκθεση τη υπάρξης αρμοστία του ΟΗΕ. Η Μεσόγειο γίνεται ένα τεράστιο νεκροταφείο. Μια θάλασσα θανάτου για άτομα τα οποία περιμένουν ανώνυμα και τους ενώνει μονάχα η προσπάθειά τους να διασωθούν και να σώσουν τις, τις ζωές των παιδιών τους και να βρουν μια ζωή ελευθερίας και ειρήνης. Η Προεδρία τώρα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία του Χαρτούμ, η οποία περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια σειρά καθεστώτων στο κέρας της Αφρικής με στόχο να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια δεν θα γίνονται από τις μετανάστες. Εμείς χαιρετίζουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να επιτύχει κάτι τέτοιο. <clears throat> δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να φανταστούμε καν ότι καθεστώτα όπως αυτά του κέρδους Αφρικής τα οποία καταπιέζουν τους πολίτες τους σε τέτοιο βαθμό ώστε προσπαθούν αυτοί να διαφύγουν θα επιτύχουν αυτό το στόχο. Το Σουδάν, η Σομαλία και η δικτατορία στην Ερυθρέα η οποία είναι απόλυτα ανελέητη έναντι των πολιτών της και η οποία φυλακίζει τους πολίτες της χωρίς αποχρόντα λόγο. Και υπάρχουν άτομα που μένουν στις φυλακές για χρόνια χωρίς τη δυνατότητα να έλθουν ποτέ ενώπιον ενός δικαστηρίου. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα και το κάνω αυτό κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να καθορίσει σαφώς τον δικό της ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε στη συνεργασία δικρατοριών για να βρούμε λύσεις στα προβλήματα μετανάστευσης. Τακ. Τακ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ε, έχετε μια μπλε κάρτα όμως από τον κύριο Κάρβερ. Τη δέχεστε την ερώτηση. Παρακαλώ, κύριος Κάρβερ. Ευχαριστώ, συνάδελφε, που δέχεστε την ερώτησή μου. Άκουσα τα σχόλιά σας ως προς τις δικτατορίες. Θα συμφωνήσετε ε, με τον αποτροπιασμό μου ότι μία από αυτές ήταν η Αιθιοπία που είχε ένα τρομερό καθεστώς του ε, Προέδρου Μεγκίστου ε, που ζούσε σε πολιτική, σε πολυτελή ανακτορά και ζήτησε και άσυλο στο Ζιμπάμπουε συμφωνείτε να εκδοθεί στην Αιθιοπία μαγιστού, Μαγκίστου ε, γιατί ε, κατηγορείται για γενοκτονία εκεί και έχει μάλιστα καταδικαστεί η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που πρέπει τώρα να κάνουμε είναι να πούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθούμε οι δικτάτορες να ορίζουν τους κανόνες για μας, τις ευρωπαϊκές ελεύθερες δημοκρατίες, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι η δική μας πολίτης, ο δικός μας πολίτης, ο Δαβίδης Σάκ, πούμε, που κρατείται πάνω από 4.000 ημέρες στην Ερυθρέα, που είναι από τα πιο σκληρά δικτατορικά καθεστώτα στον κόσμο. Με αυτούς θα πάμε να συνεργαστούμε. Εμείς θα τους εμπιστευτούμε ότι θα ε, βαστούν και θα ε, σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θα πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι αμφιβάλλω πολύ γι' αυτό. Είναι δική μας ευθύνη και δεν μπορούμε ποτέ να το αναθέτουμε ε, σε τέτοια καθεστώτα στη διαδικασία της χαρτού. Την χαιρετίζομαι, αλλά φοβάμαι ότι θα αποτύχει από χέρι γιατί δεν μπορούμε να έχουμε διγλωσία, μία γλώσσα και μία σαφή φωνή πρέπει να έχουμε για την ελευθερία του λόγου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ε, ακολουθεί από την Ενωτική Αριστερά η κυρία Βερζιά. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία του Χαρτούμ έχει παρακαλώ ως στόχο να εξομαλύνει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του κέρατος της Αφρικής. Φυσιολογικό και μπανάλ. Είναι ένας διάλογος με δικτατορίες που παραβιάζουν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο κόσμος τους ξενιτεύεται για να ξεφύγει από την καταστολή. Η Ιταλική Προεδρία μεταξύ άλλων θέλει, λέει, να ενθαρρύνει την πλήρη ένταξη της Ερυθρέας ως χώρας κλειδί στη διεθνή κοινότητα. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να βάλετε τα θεμέλια μιας πολιτικής συνεργασίας ουσιαστικής, λέτε, με αυτές τις χώρες προέλευση. Το ίδιο μας είπε και το Συμβούλιο. Μάλιστα μας είπατε στην Επιτροπή ότι αν το πρόβλημα ήταν το όνομα της διαδικασίας να το αλλάξουμε. Όχι, είναι ένα θέμα ε, χωρών προέλευση, διέλευση και θα πρέπει να αποφύγουμε να ε, φεύγουν από τις χώρες τους οι μετανάστες και να μένουν ατιμόρυτοι οι κυβερνώντες. Τι διάλογο μπορεί να κάνουμε με τέτοιες κυβερνήσεις που επιζητούν τη διεθνή αναγνώριση και εσείς αυτό κάνετε. Επαναλαμβάνω, το λέω και ξανά και ξανά, συμμετέχουν σε όλα τα λαθρεμπόρια στην περιοχή. Πώς μπορείτε να μας λέτε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στην καρδιά αυτής της διαδικασίας και παραμένουν προτεραιότητα. Πώς μπορεί να μας λέτε ότι έτσι θα σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουλευτά. Και τώρα από τους Πρασίνους το λόγο έχει η κυρία ε, Ιούντι της Αρχεντίνη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περίεργη συνάντηση θα ήταν αυτή στη Ρώμη με εκπροσώπους του Σουδάν, του Νοτίου Σουδάν, της Αιγύπτου, Αιθιοπία, Ερυθρέα. Η Λιβύα που είναι, σας ξέφυγε. Δεν τη βλέπω στον κατάλογο. Και στη Λιβύη ποιον θα ζητήσουμε, από ποιον να εκπροσωπεί την κυβέρνηση της χώρας. Ε, θυμούμε πριν από λίγα χρόνια μια συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο για τον deal, τη συμφωνία που είχε κάνει με τη Λιβύη η Ιταλική κυβέρνηση για να τους ε, φιλοξενεί η Λιβύη. Και θυμάμαι τότε την κυρία Μάλστρομ, προκάτοχο του κυρίου Αβραμόπουλου, που έπρεπε να πάει στη Λιβύη για να φροντίσει 250 πολίτες Ερυθρέας που είχαν ε, αποσταλεί πίσω από την Ιταλία να μην τους στείλουν στην Ερυθρέα γιατί θα τους σκότωναν καθίσαμε εδώ για να συζητήσουμε με το πώς θα κρατάτε τους μετανάστες σπίτι τους, με ε, καθεστώτα που αφανίζουν, σκοτώνουν ανθρώπους. Τους σκοτώνουν κανονικά και παίρνουν και ε, κονδύλια από την επίσημη αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτή η διαδικασία του Χαρτούμ δεν είναι μόνο το όνομα. Και πώς έτσι και μπορούμε να αρχίσουμε μια διαδικασία στην πρωτεύουσα του Σουδάν. Δεν είναι το όνομα. Είναι με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία και πώς ε, ε, θα ε, σπρώχνει πίσω μετανάστες η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το μαδία της αναπτυξιακής βοήθειας ενώ θα τα έχει κάνει πλακάκια με δικτατορίες. Ευχαριστώ πολύ. Από την ομάδα του τώρα το λόγο έχει ο κύριος James Carver. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε ανθρώπους απελπισμένους και γενναίους να ξεφύγουν από τον δρόμο ε, της άκρεας φτώχειας και των σειράξεων. Οποιαδήποτε τέτοια βοήθεια όμως θα πρέπει να είναι εφικτή, εφαρμόσιμη και προς το συμφέρον όλων και να μην ενθαρρύνουμε μια κακή κατάσταση να χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της μετανάστευσης αν θέλουμε να αποθαρρύνουμε τον κόσμο να πηγαίνει να πνίγεται στη Μεσόγειο με σαπιοκάραβα. Αλλά η διεθνής κοινότητα και τα κράτη ε, τα έθνη δεν ε, το πράττουν. 500 εκατομμύρια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί ε, να αναλάβει όλους τους μετανάστες. Στο Σουδάν, στο νότιο Σουδάν, στη Σομαλία, Ερυθρέα, Αιθιοπία, Κένια και Ουγγάντα είναι 4,3 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι θα πρέπει να δούμε πώς έχει αυτή η διαδικασία ε, και τι επιπτώσεις έχουν άλλες πολιτικές της Ένωσης στην Αφρική, η κοινή γεωργική πολιτική. Δεν είναι μόνο σπατάλη για το Βρετανό φορολογούμενο, αλλά στέλνει στην αφρικανική οικονομία επιδοτούμενα γεωργικά προϊόντα και τη βυθίζει στη φτώχεια. Ε, να μην μιλήσω για την αλία στη Σομαλία, πώς έχουμε καταστρέψει τον κόσμο και πώς τους σωθούμε στη φτώχεια ή στην πειρατεία ή στο εμπόριο που είναι πολύ υψηλή η φραγμή που βάζουμε οι δασμολογικοί και εμποδίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ανεπανόρθωτες ζημίες σε όλη την Αφρική χρειάζεται αξιοπρέπεια και σεβασμό στις σχέσεις μας. Θα πρέπει να αρθούν οι φραγμοί που έχουν επιβάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσουμε το κακό στη ρίζα του. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της διεθνούς κοινότητας. Γιατί συνεχίζει να αντιτίθεται στην αναγνώριση της Σομαλιλάνδης. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται το κέρας της Αφρικής είναι χώρες σταθερές, ασφαλείς που να μπορούν να εξασφαλίζουν ζωή για τους πολίτες τους μόνο εάν αναδείξουμε την επιτυχία του σαξτές του Σομάλιλαντ θα βοηθήσουμε την περιοχή. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Μην τους δίνουμε δώρα. Δώστε ε, όλη την Αφρική ελπίδα και οι άνθρωποι θα κανονίσουν τις ζωές τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει από τους μία εγγεγραμμένους ο κύριος Συναδεινός. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, 200.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι νέοι, μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια διωκόμενοι από το καθεστώ τη χώρα του. Οικονομικοί μετανάστε στα όρια τη φτώχεια, άνεργοι, χωρί αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αφήνοντα πίσω κατοικίε υπό τον κίνδυνο κατάσχεση από τι τράπεζε. Αυτή η χώρα δεν είναι το Σουδάν, ούτε ανήκει στην Υποσαχάρη Αφρική. Είναι η Ελλάδα, χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, δυστυχώ έχει πολλά κοινά με τη χώρα που σκέφτεστε να βοηθήσετε σήμερα. Αυτοί οι 200.000 Έλληνε που μετανάστευσαν λόγω της κρίσης είναι νέοι επιστήμονες έως 40 ετών. Φωτεινά μυαλά με όρεξη για εργασία χωρίς όμως μένο στην πατρίδα μου την Ελλάδα. Σίγουρα η μετανάστευση από την Αφρική στις χώρες της Ευρώπης αποτελεί μείζον πρόβλημα. Εμείς το ξέρουμε καλύτερα διότι το αντιμετωπίζουμε μόνοι μας έχοντας απέναντί μας την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας επιβάλλει να δεχόμαστε στη χώρα μας παράνομους μετανάστες όπως ορίζει η συνθήκη του Δουβλίνο 2. Είναι όμως ανοησία να χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα περιορισμού των μεταναστών από την αφρική όταν δεν ενδιαφέρεται να περιορίσει την εσωτερική μετανάστευση που προκλήθηκε λόγω των κακών πολιτικών τη. η εσωτερική μεταναστευτική ροή αποδεικνύει ότι οι χώρε του εύρου του βορρά καταδικάζοντα τι χώρε του νότου σε οικονομικό μαρασμό και εξαθλίωση προσελκύουν το πιο αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λένας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χρειάζεται διαρθρωτική προσέγγιση της μετανάστευσης, αυτό το έχουμε καταλάβει όλα. Και θα πρέπει να είναι σφαιρική, ολιστική αντιμετώπιση της μετανάστευσης και αυτό το έχουμε καταλάβει. Και το λέμε και στο ψηφίσμά μας ε, χρειάζεται να συντονίζεται περισσότερο η εσωτερική πολιτική της Ένωσης με την εξωτερική της πολιτική. Και είναι καλό που κοιτάει ο Επίτροπος και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης και συνεργάζεται με τρίτες χώρες. Τώρα που συζητούμε για τη διαδικασία του χαρτού, αν κοιτάξετε το γεωγραφικό χάρτη της Αφρικής και τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, μεταξύ της Ισίας και Αιγύπτου υπάρχει ε, μια λευκή ή μαύρη τρύπα και αυτή είναι η Λιβύη ε, που δεν εγγράφεται σε αυτή τη διαδικασία ή τη διαδικασία Ραμπάτ. Ε, η Λιβύη είναι μια χώρα διέλευσης πάρα πολλών ανθρώπων που φτάνουν στη Μεσόγειο. Τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί χωρίς ε, να ε, δείτε τι συμβαίνει στη Λιβύη. Πώς θα το λύσετε αυτό στα πλαίσια της διαδικασίας Χαρτούμ. Ε, Σας ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ραντζουλίτσα. Ένοπλες σειράξει, έλλειψη οικονομικών προπτικών, φυσικές καταστροφές, θεομηνίες αναγκάζουν τον κόσμο να, φεύγουν από τα σπίτια τους, από το κέρα της Αφρικής και να ξεκινούν επικίνδυνες ε, πορείες, διαδρομές ε, ανάμεσα σε διάφορες χώρες για να προσπαθήσουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Στη διάρκεια του ταξιδιού οι προσωπικέ του επίδεση ε, για ευτυχία συχνά καταστρέφονται από το οργανωμένο έγκλημα, από τους λαθρέμπορες, δουλέμπορες, έλλειψη νερού και τροφίμων στη διάρκεια του ταξιδιού. Και όταν φτάσουν, αν φτάσουν στην Ευρώπη, καλωσορίζονται από το ρασισμό, την εκμετάλλευση και τον αποκλεισμό. Αν όμω επιτείνουμε τι προσπάθειέ μα και τι πολιτικέ μα, θα αλλάξουμε τι ζωέ εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι αποφάσει μα θα βελτιώσουν την ευημερία και τι συνθήκε διαβίωση των ε, μεταναστών. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι ρίζε τη μετανάστευση, αν στηρίξουμε κυβερνήσει, με διάφορου οργανισμού αλλά και πολίτε για να αναπτύξουν καλή διακυβέρνηση και να δημιουργήσουν μια πιο ευημερή κοινωνία, ίσως τελικά η μετανάστευση θα είναι μια ελεύθερη επιλογή. Να θυμίσουμε δε ότι πόσο έχουμε κερδίσει από διάφορους μετανάστες που έχουν σε καλά ενσωματωθεί στις χώρες ε, προέλευσης αλλά και στις χώρες προορισμού. Η σωστά διαχειριζόμενη μετανάστευση μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση την οικονομική της χώρας μέσω των εμβασμάτων που γίνονται προς τα εκεί. Οι νέοι μπορεί να αποκτήσουν ε, ε, νέες γνώσεις και δεξιότητες αν μπορέσουμε να καταστήσουμε σαφές μέσα στο δικό μας το μυαλό αλλά και ευρύτερα πως υπάρχει αναμφίβολα θετική σύνδεση ανάμεσα στη μετανάστευση και την ανάπτυξη τότε θα πάψει να είναι πρόβλημα η μετανάστευση και θα είναι τμήμα της λύσης. Ευτυχώς αυτή η σύνδεση ε, ε, ε, κατέστησε αφής που ε, στην, στα, στις δηλώσεις του Συμβουλίου την περασμένη φορά για την αναπτυξιακή συνεργασία. Ελπίζω να δούμε πώς η Κομισιόν θα θέσει σε εφαρμογή αυτά τα πορίσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, υπάρχει μπλε κάρτα για σας από τον κύριο Κάρβερ και από την κυρία Σπινέλη. Δέχεστε αυτές τις δύο μπλε κάρτες. Ε, ναι, η κυρία Σπινέλη θα μιλήσει πρώτη. Συνάδελφε, εδώ βρίσκομαι. Εδώ, εδώ. Συνάδελφε, συμφωνώ πως χρειάζεται να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, των προβλημάτων, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν λέτε πως χρειάζεται να βοηθηθούν και να στηριχθούν οι κυβερνήσεις ε, των χωρών από όπου έρχονται οι μετανάστες και ότι αυτό είναι μία από τις ρίζες του προβλήματος, δηλαδή τα κράτη των προέλευσης των μεταναστών, εσείς έχετε υπόψη σας από τι χώρες φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Τους πολέμους, την πείνα, τις δικτατορίες, τις φρικτές, τις Από εκεί που φεύγουν αυτοί οι μετανάστες, γιατί δεν έρχονται γιατί δεν υπάρχει μόνο αρκετή ανάπτυξη. Έρχονται γιατί διαφορετικά θα βρεθούν στη φυλακή. Με γνωρίζω πολύ καλά για ποιες χώρες μιλώ. Όπω γνωρίζετε, υπάρχουν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάποιες από αυτές τις χώρες επίσης και όλα αυτά τα προγράμματα θα έπρεπε να να, να περιέχουν κάποιους όρους από πλευρά μας ώστε οι κυβερνήσεις αυτές να αναγκαστούν να εφαρμόσουν περισσότερη ε, νομοθεσία και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία αλλά και αν είναι δυνατόν να προωθήσουν μια οικονομία της αγοράς. Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές ώστε να δώσουν, στους προσφέρουν στους πολίτες τους λόγους για να μείνουν στη χώρα τους. Ο κύριος Κάρβερ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που δεχτήκατε την μπλε κάρτα συνάδελφε. Συνάδελφε, εσείς μοιράζεστε το πάθος μου για μια ανεξάρτητη Σομαλιλάνδη που θα αναγνωριστεί στον ΟΗΕ και από τη διεθνή κοινότητα και συμφωνεί μαζί μου ότι ίσως είναι λιγότερο πιθανή και λιγότερο βιώσιμη η επιλογή για την αναγνώριση του Νοτιού Σουδάν που είναι η τελευταία χώρα που αναγνώρισε ο ΙΕ. Λοιπόν, δέχεστε ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η Σομαλιλάνδη. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το σημερινό θέμα. Ξέρετε ότι όλες οι χώρες υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή τη Σομαλία που έχει διεθνώς αναγνωριστεί. Αλλά και πάλι να σας πω ότι το ερώτημά σας είναι εκτός θέματος. Ε, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Ντεσαρνές έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχουμε πράγματι ανάγκη να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό στην Ευρώπη. Έχουμε ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική κοινή πολιτική μετανάστευση, κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα στην Ευρώπη, γιατί τα θέματα μετανάστευση παραμένουν στο εθνικό επίπεδο με τα προβλήματα τα οποία αυτό συμπαρομαρτεί. Πρέπει να υπάρξει μια εταιρική σχέση με την Αφρική, λέτε. Εντάξει, είναι πολύ καλό να έχουμε επαφή με κάποιες κυβερνήσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάποια περισσότερη επαφή με την αντιπολίτευση, την κοινωνία των πολιτών, της ΜΚΟ. Χρειαζόμαστε μια ουσιαστική εταιρική σχέση με την Αφρική. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα αυτό, αυτό είναι κεφαλαιόδες. Θα πρέπει να δράσουμε υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης και να το κάνουμε <clears throat> με έναν τρόπο ο οποίος είναι διαρθρωμένος. Να σταματήσουμε να στέλνουμε προϊόντα τα οποία επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία καταστρέφουν την τοπική γεωργία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αποκομίσουν μια αυτάρκεια στον τροφιμικό τομέα. Είναι μια τέτοια μεταρρύθμιση που χρειάζεται. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να εργαστεί με, όλους τους, ε, με όλες τις χώρες της Αφρικής να αντιμετωπίσουμε την ε, λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι οποίοι υφίστανται πιέσει στη χώρα τους και καταδιώξει να μην μπορούν να έρθουν σε εμά για να ζητήσουν άσυλο και να πρέπει να περιοριστούν σε μια πρεσβεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα προέλευσης. Θα πρέπει λοιπόν να εναρμονιστεί το δίκαιο σε σχέση με το άσυλο. Θα πρέπει να υπάρξουν νόμιμες ποσοστώσει μετανάστευση και να υπάρχει καλύτερο έλεγχο στα σύνορά μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρος. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη έχει το λόγο τώρα. Ένα λεπτό. Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος ενός σωρό οργανώσεων, ενώσεων που, κατα... που, που καταγγέλουν την ε, διαδικασία του χαρτόμα και την... Ε, τα όσα γίνονται στα σύνορα που γίνονται αποθήσεις αντίθετες με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 30% από τους 350.000 ε, κόσμο που έχουν έρθει στην Ιταλία είναι από την Ερυθρέα. Είδαμε να υπάρχουν καταστροφές, ε, ακόμα και εξαγωγή των μεταναστών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και αυτό ακόμα ε, οδηγεί σε καταστροφές και απάτες. Ε, η διαδικασία της Χαρτούν περιγράφεται από την Ιταλική Προεδρία ως μια, ένα ιστορικό άλμα ποιοτικό. Εμεί ε, στην ουσία κάνουμε νέε συμφωνίε με τις χώρε διέλευση για να σταματήσουμε τις αναχωρήσεις, για να μην χρειάζεται να δοθεί το δικαίωμα ασύλου που ήδη δεν είναι εγγυημένο ούτε και επί τη βάση των πιο περιοριστικών προβλέψεων της Σύμβασης της Γενέβης. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Φεράρα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε διαδικασία της χαρτών προκύπτουν ε, υποκρισίες για μια δύσκολη συνεργασία που μπορεί να βασιστεί μόνο σε ένα σε μια, ένα πολύ ευαίσθητο και ευάλωτο ε, καράβι. φαίνεται να είναι λυπής και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από τη μια πλευρά λέτε ότι θέλετε να αναχαιτήσετε το δουλεμπόριο και τις δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων που εκμεταλλεύονται τους, τους μετανάστες. Από την άλλη πλευρά έχουμε καθεστώτα δικτατορικά, αιματηρά ε, ε, σκεφτείτε μόνο την υπόθεση, της, ε, την περίπτωση της Ερυθρέας με, με πολύ σκληρή δικτατορία, με χιλιάδες κόσμο στις φυλακές ή την ε, περίπτωση του Σουδάνου όπου εδώ και δεκαδίες γίνονται γενοκτονίες και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και άλλες κυβερνήσεις όπως αυτή της Αιθιοπίας ή της Αιγύπτου έχουν αποδείξει ότι δεν λάμπουν όσον αφορά τα δικαιώματα τα ανθρώπινα. Και για τη Λιβύη ποτέ δεν κύρωσε τη σύμβαση της Γενέβης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, ωστόσο δήλωσε ότι θέλει να προωθήσει συνεργασία σε θέματα ασύλου και διεθνού προστασία επί τη βάση των αρχών του διεθνού δικαίου, αναφερόμενη στην ίδια αυτή σύμβαση. Η Λιβύη, μια από τι χώρε όπου συγκεντρώνονται χιλιάδε μετανάστε και που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη, ούτε καν συμμετείχε στη συνάντηση τη Ρώμη τη 28 Νοεμβρίου, όπου υπογράφηκε η κοινή δήλωση τη για τη διαδικασία τη Χαρτούμ, έτσι ώστε να υλοποιηθούν εκτό ε, των Ευρωπαϊκών Συνόρων κέντρα υποδοχή. Εδώ θα εξετάζονται υποθέσεις των ετούντων άσυλο. Αντί να καταπολεμηθούν τα αίτια της μετανάστευσης, στόχος είναι να βρεθούν οι συμφωνίες για το πώς θα σταματήσουμε τους μετανάστες πριν καν βάλουν το πόδι τους στην Ευρώπη. Ξεχνώντας ε, την εμπειρία ανάμεσα στον Κατάφη και τον Περλουσκόνη. Ξεχνάμε ότι υπάρχουν μεγάλες επίγουσες καταστάσεις ε, και ανάγκες ε, μπορεί ακριβώς αυτά τα στατόπεδα ε, υποδοχής να μετατραπούν σε γκέτο όπου δεν θα είναι καθόλου εγγυημένα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας να σταματήσει η υποκρισία. Θα πρέπει να εγγυηθούμε την ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση και την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα δικαίωμα σε άσυλο λαμβάνοντας υπόψη τους πιο ευάλωτους όπως οι ανήλικοι μετανάστες. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φρανκ Έγγελ. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στα πολωνικά ο κύριος Έγγελ. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας την κυρία Σπινέλη ότι αν εκείνη μιλά για όλους εκείνους που φεύγουν από το κέρας της Αφρικής ε, για να αποφύγουν τη φυλακή σε μια χώρα όπως η Σομαλία δεν υπάρχουν αρκετές φυλακές γιατί αυτός ο κόσμος δεν φεύγει από τη φυλακή αλλά φεύγει από την έλλειψη κράτους ενώ εμείς ε, παριστάνουμε πως εξακολουθεί να υπάρχει κράτος εκεί ενώ η Σομαλία δεν υπάρχει πλέον. Πράγμα το οποίο με οδηγεί σε κάτι που ο συνάδελφο Κάρβερ μάλλον θα εκτιμήσει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για τη Σομαλιλάνδη και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό και γρήγορα γιατί είναι περίπου η μόνη περιοχή σε ολόκληρη την περιφέρεια που όχι μόνο δημοκρατικά έχει συσταθεί αλλά και που μπορεί να αποτελέσει και ένα καταφύγιο για μεγάλο αριθμό ανθρώπων γύρω από εκεί που δεν έχουν που να φύγουν και αυτό ήταν το πιο ασφαλές καταφύγιο που θα μπορούσαν να φτάσουν, το πιο κοντινό. Και τέλος για να κλείσω και να πω κάτι στην Κομισιόν. Πήραμε αυτό το όνομα για αυτή τη δικασία από μια πρωτοβουλία της Αφρικανικής Ένωσης. Στο όνομα της συνοχής των πολιτικών που συχνά αναφέρεται και για το οποίο ε, αισθάνομαι δεσμευμένος, θα πρέπει όντως να προσπαθήσουμε και να ακολουθήσουμε τις πρωτοβουλίες της ίδιας Αφρικανικής Ένωσης, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε φαινόμενα που θέλουμε να περιορίσουμε. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αν θέλουμε και πρέπει να συνομιλήσουμε με δικτάτορες, ίσως να μην είναι το πιο ευχάριστο πράγμα να κάνει κανείς, αλλά ε, ίσως να είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε για να επιτύχουμε ένα στόχο. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η Άννα Γκόμες για ένα λεπτό. Έχουμε δικτατορίες οι οποίες ε, καταπιέζουν τους λαούς τους και δεν σέβονται τα δικαιώματα των μεταναστών, δεν σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών, όλων αυτών οι οποίοι κινδυνεύουν τη ζωή τους και τους εκμεταλλεύονται οι διακινητές. Οι κυβερνήσεις αυτές οι οποίες είναι εγκληματικές από την Ερυθρέα που καταπιέζουν το λαό τους, οι Όλοι αυτοί είναι μηχανές παραγωγής μεταναστών. Τα καθεστώτα αυτά τα καταπιεστικά είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο χιλιάδες από τους πολίτες τους προσπαθούν να φύγουν για να διασώσουν τη ζωή τους. Εάν η Ευρώπη θέλει να σταματήσει τη μετανάστευση, πρέπει να δώσει στους λαούς αυτούς τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από τις καταπιεστικές αυτές δικτατορίες, αντί να πληρώνουν αυτές οι δικτατορίες για να διατηρούν φυλακές στο έδαφος τους και με διαδικασίες όπως αυτή του Χαρτούμ που είναι καταδικασμένη στην αποτυχία. Και είναι σαν τις προσπάθειες που κάνανε η Ιταλία και η Ευρώπη για να έχουν τέτοια κέντρα κράτησης στην Λιβύη. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να σταματήσει την κατάσταση αυτή που επικρατεί εφηλίου πολέμου στην Συρία, να σταματήσει η αντιπαράθεση Ισραήλ-Παλαιστίνης, η κατάσταση στη Γάσα που και αυτή παράγει ε, <clears throat> μετανάστες. Είναι λοιπόν η κτρή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Λιβύης γιατί από την χώρα αυτή φεύγουν οι περισσότεροι μετανάστες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το κέρας της Αφρικής. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Μπιλμπάου Μπι Μπαράντικα έχει το λόγο. Για τρία λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ευρωπαϊκές χώρε που έχουν δεσμευτεί να ξεκινήσουν τη διαδικασία του χαρτούμ, ιδίω αυτέ, οι οποίε είναι πιο μακριά από τι ε, σχεδίες και τι ταγωδίε τη Μεσογείου, θα πρέπει να αναλάβουν ένα πρόβλημα που, ισχύει για όλου. Ελπίζω ότι η συνάντηση τη Ρώμη 28 Σεπτεμβρίου και οι δράσει τη κυρία Μογκερίνη θα μπορέσουν να βοηθήσουν να αναρθώσουν μια πολιτική που να βασίζεται περισσότερο στην αλληλεγγύη, στη συνεργασία και στην σωστή αντιμετώπιση. Έχουν συμμετάσχει 38 χώρε, οι οποίε ε, συνεργάζονται για την ε, ανάπτυξη και τη συνεργασία, για την ε, ειρήνευση, για την σταθεροποίηση τη δημοκρατία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να μετακινήσουμε το δράμα από τις ακτές της Μεσογείου στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερο. Ο Ντένις Μουκουέβε, το βραχυδίο Σαχαρόφ, μας εξήγησε πάρα πολύ σαφώς τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί τόσο κόσμο να εγκαταλείψει τι αιστείες του. Πολλές φορές είναι οι πόλεμοι οι οποίοι προκύπτουν από <clears throat> εμπορικές ε, εμπορικά συμφέροντα τα οποία έχουν να κάνουν με τη θέληση ενός τυράννου μονάχα. Μιλώντας για την περίπτωση του Αναστάσιου Σωμός, ο πρώτο Ρούσβελτ είπε. Δεν θα είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο θα πω από πολιτική άποψη. Είπε, είναι ένας τύρανος, αλλά είναι ο δικός μας τύρανος. Θα πρέπει να νιώσουμε ντροπή όταν βλέπουμε τους ηγέτες μας να φωτογραφίζουν μαζί με τέτοιους δικτάτορες. Θα πρέπει να κάνουμε ένα κατάλογο των ωφελουμένων από αυτές τις δικτατορίες και να εμποδίσουμε να συνεχίσει αυτό το αίμα, αυτή η καταστροφή. Γιατί ο τύρανος είναι πάντα τύρανος. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ε, η ε, επόμενη ομιλήτρια. κυρία Πιόρκ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι ε, σιγά σιγά χτίζουμε πετραδάκι πετραδάκι το φρούριο Ευρώπη και τώρα φτιάχνουμε και μία τάφρο γύρω γύρω. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Ε, χρήματα από την αναπτυξιακή βοήθεια θα πάνε σε αυτό το σκοπό. Είναι πραγματικά διασπάθηση. Ε, προσπαθούμε να αποθήσουμε μετανάστες, πρόσφυγες. Ε, σκεφτείτε ποια είναι η αφετηρία. Κανονικά εμείς θα πρέπει να ε, αυξήσουμε τις πιθανότητες επιβίωσης των ανθρώπων όταν φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες. Ε, θα ήταν τελείως διαφορετική η πρωτοβουλία αν είχαμε αυτό στο μυαλό μας όταν ξεκινούσε. Άκουσα τον κύριο Έγγελ και άλλους από τη δεξιά. Αν τα πράγματα πάνε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα πάρουμε άλλες αποφάσεις. Ελεύθερο εμπόριο, έλεγχο των μεταναστευτικών ρευμάτων, συνεργασία με δικτάτορες και όλα αυτά θα είναι στο βωμό ε, της προστασίας των ανθρώπων. Άσυλο ζητάει ο κόσμος. Αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαριάννα Πέτυρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. 40.000 περίπου μετανάστες και εκτοπισμένοι ήρθαν το 2013 στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό ε, Μετανάστευσης, πάνω από 3.000 φέτος έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο. Δυστυχώς το 2014 έτσι έγινε το πιο ε, θανατηφόρο έτος ε, στη Μεσόγειο, όπου ο κόσμος πνίγηκε ε, στις θύρες της Ευρώπης. Και υπήρξαν και άλλοι θάνατοι από την πείνα, όχι από πνιγμό. Οι περισσότεροι ερχόνται από την Ανατολική Αφρική. Η διαδικασία του Χαρτούμ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χαιρετήσουμε, διότι αποτελεί ένα πλαίσιο διαλόγου μεταξύ Αφρική και Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε αυτή τη διακίνηση ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να έχουμε συμμαχίες και συνασπισμούς ή βοήθειες γενικά και αόριστα. Ούτε μας ενδιαφέρει να ε, ξεπλύνουν τη συνείδησή τους οι πολιτικοί με το χρήμα ε, γιατί επεμπόλησαν τις ευθύνες τους. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ε, ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος μας τα είπε αυτά εδώ της προάλλης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η Ευρώπη, η Μεσόγειος να γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο. Ε, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την μετανάστευση θα λυθούν μόνο εφόσον η Ευρώπη ξέρει ποια είναι η πολιτιστική της ταυτότητα και υιοθετήσει εκείνη την νομοθεσία για να προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και να υποδέχεται και τους ε, μετανάστες. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα, το κακό στη ρίζα του και όχι στις συνέπειες μόνο. Η κυρία Κιέγκε για ένα λεπτό και μισό. Ε, ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τεράστια ε, ε, ροή μεταναστών αντιμετωπίζει η Ευρώπη και αυτό αναγκάζει την υιοθέτηση ε, μηχανισμών πολυμερού συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών μέσα από προτάσεις που θα έπρεπε να είναι βιώσιμες και σταθερές. Μία χώρα δεν μπορεί μόνη της να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Θα πρέπει να βασιστεί ένα σχέδιο σε διάλογο και κοινού πόρους αλλά κυρίως στην πολιτική βούληση με στόχο να σωθούν ε, χιλιάδες ε, μεταναστών από τους ε, δρόμους του θανάτου. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ροές μεταναστών μέχρι ότου δεν θέσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και κυρίως σε μια παγκόσμια, σε μια καθολική μάλλον και ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση. Γι' αυτό και εκφράζω επιφυλάξεις όσον αφορά το τελευταίο πόρισμα που περιγράφεται στην διαδικασία της Χαρτούμα. Αναφέρομαι στη δυνατότητα τα δημιουργία ε, στρατοπέδων προσφύγων ως ε, ε, κέντρα υποδοχής ή κράτησης. Τον άσυλο θα πρέπει πάντα να λέει να συνοδεύεται από μια διαδικασία επαλήθευσης της, των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως της στήρησης όλων των διεθνών συμβάσεων. Ποιος θα είναι ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου. Θυμίζω τις συμφωνίες με τη Λιβύη από πλευράς της Ιταλικής κυβέρνησης και δεν θέλουμε να υπάρξει παρόμοια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα γνωρίζουμε όλοι πω ορίστηκε η κυβέρνηση του Γκαντάφη. Ευχαριστούμε. Χωάν Φερνάντο Λόπετ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, η διαδικασία του χαρτού είναι ε, κάτι που ε, έχει θλιβερά επεισόδια και λυπούμαστε. Λαμπεντούζα, 400 νεκροί. Κάθε φορά επιγόντως θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους διαλόγου και συνεργασίας με χώρες προέλευσης, διέλευσης ή προορισμού. Ε, αυτού ε, του λαθρεμπορίου, της διακίνησης ανθρώπων με τραγικές συνέπειες. Ο στόχος θα πρέπει να ίδιος και στο κέρα της Αφρικής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ούτε στιγμή ότι όταν μιλάμε για Αιθιοπία, Σομαλία, Ερυθρέα, πρόκειται για χώρες που πολύ συχνά είναι χώρες ε, χρεοκοπημένες, αποτυχημένες, χωρίς διοίκηση, χωρίς σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς καμία εγγύηση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αυτή τη συνεργασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συνεχίσει να τηρεί τα ίδια της πρότυπα για τα θεμελιώδη δικαιώματα να αποτρέψουμε τη διακίνηση ανθρώπων, ναι. Το λαθρεμπόριο, ναι. Να εξασφαλιστεί ο διάλογος, ναι. Αλλά πάντα με τη μεγαλύτερη απέτηση κάθε ευρώ που θα ε, δαπανάτε εκεί για να ε, αντιμετωπιστούν ε, οι τεράστιες αδικίες να μας οδηγεί ένα βήμα μπρο για τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πιο ευαλώτων που είναι οι γυναίκες, οι ανήλικοι που πέφτουν θύματα σε αυτό το λαθρεμπόριο με τραγικές συνέπειες που κάθε φορά ξανά και ξανά θρυνούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Κριστίν Γοβονταλών για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια ε, καθολική και πλήρης ε, ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση απαιτεί μόνιμο διάλογο με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Η διαδικασία Χαρτούμ με το κέρας της Αφρικής συμμετέχει σε αυτό. Τα συμβαλόμενα μέρη βάζουν την κορφή των προτεραιοτήτων, την καταπολέμηση της διακίνησης των δικτύων και ε, τα αίτια. Προσοχή όμως αυτή η φιλοδοξία να μην είναι πρόφαση για να υψωθούν νέα εμπόδια στη μετανάστευση. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να φύγει από τη χώρα του για να βρει καλύτερη μοίρα ή να ζητήσει άσυλο θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη για να τερματιστεί η τραγωδία στη Μεσόγειο. Η συζήτηση για την νόμιμη μετανάστευση που εμφανίζεται ως επόμενη ε, φάση του διαλόγου ε, Χαρτούμ θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα και για να υπάρξει πραγματική προτιθέμενη αξία δεν θα πρέπει να είναι μόνο δήλωση προθέσεων η διαδικασία. Τα λόγια θα πρέπει να συνοδεύονται από έργα συγκεκριμένα για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ετούντων άσυλων και των μεταναστών. Ωστόσο, όλα αυτά θα γίνουν ε, σε εθελούσια βάση. Δεν υπάρχει καμία νομική δέσμευση σε ε, σχέση με ε, το διεθνές δίκαιο. Πού είναι η προστιθέμενη αξία, πού είναι η αναγκαστική ισχύ και πώς θα εξασφαλίσουμε την προστασία των μεταναστών και την πλήρη, τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων του δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Βουλευτά. Και Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Δύο βουλευτές έχουν ζητήσει. Ο κύριος Μαριάς πρώτο. Προκειμένου να περιοριστούν οι μεταναστευτικές τροές από τις χώρες που ανήκουν στο κέρας της Αφρικής, πρέπει να εκλείψουν οι βασικές αιτίε που προκαλούν το πρόβλημα αυτό, που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές. Και φυσικά το πρώτο και βασικό είναι να ανατραπούν τα δικτατορικά καθεστώτα τα οποία υπάρχουν στις χώρες που ανήκουν στο κέρας της Αφρικής να επανέλθει και να στηριχθεί εκεί η δημοκρατία να σταματήσουν οι διώξεις να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. δεύτερον πρέπει να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή γιατί όσο έχουμε μια εμπόλεμη κατάσταση σε διάφορα σημεία δημιουργούνται προβλήματα και προφανώς οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν πρέπει να σώσουν τις ζωές τους. στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει οικονομική στήριξη από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης για να αναπτυχθούν οι περιοχές αυτές. να χτυπηθούν βεβαίω τα δουλεμπορικά δίκτυα και κυκλώματα. να καταργηθεί τέλος το δουβλίνο τρία το οποίο μετατρέπει τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου σε αποθήκη ψυχών καθώς εκεί εγκλωβίζονται χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες. και τέλος να γίνει αυτό το οποίο είπατε να διαμορφωθεί συνολική αντιμετώπιση και προσέγγιση στο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. ευχαριστώ. Ε, ε, και τώρα ο κύριος Ντομπάς και τελευταίος. Ε, ε, ευχαριστώ. Αγαπητοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Κομισιόν, εγώ θέλω να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο κύριος Μαριάς και να σας πω τα εξή. Άκουσα μέχρι τώρα ότι το, η μετανάστευση είναι χρήσιμη και πρέπει να την ενθαρρύνουμε και να, να, να την διοχετεύσουμε σωστά. Εμείς που είμαστε όμως άνθρωποι που ζούμε ε, στα σύνορα, Βουλγαρία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, η μετανάστευση είναι πρόβλημα και όχι ε, λύση. Αυτά τα κράτη γίνονται κατά κάποιο τρόπο στρατόπεδα προσφύγων. Ε, μαζεύεται κόσμος πολύ, σε κόσμος που δεν μπορεί να βρει δουλειά. Οι πολιτιστικές διαφορές είναι πολύ μεγάλες και σημαντικές, δεν καταφέρνουν να ενταχθούν. Είναι τεράστιο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εφόσον πρόκειται για μετανάστευση πρέπει να γνωρίζουμε σε τι οφείλεται. Να βρούμε σε τι οφείλεται στη χώρα προέλευσής του. Γι' αυτό και ρωτώ, ποιος ε, στηρίζει αυτούς τους δικτάτορες, ποιος καταστρέφει τα κράτη, ποιο κατέστρεψε τη Λιβύη, ποιο κατέστρεψε την Αίγυπτο, τη Σομαλία Ποιο κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία, πώς θα βρούμε τη λύση και πώς θα αποφύγουμε να μετατραπεί η Ευρώπη σε ένα τεράστιο στρατόπεδο προσφύγων, γιατί οι πληθυσμοί της Αφρικής ξεπερνούν το δισεκατομμύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως, τελειώσατε οι ομιλητές και τώρα το λόγο έχει ο επίτροπο Αβραμόπουλος. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί κύριοι βουλευτές. Πιστεύω ότι ένας ε, σταθερός και εξισορροπημένος διάλογος με τις χώρες του κέρατο της Αφρικής είναι απαραίτητος. Το θέμα δεν είναι κατά πόσο θα πρέπει να συνεργαστούμε ή όχι με τις χώρες αυτές, αλλά με ποιο τρόπο θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες αυτές και να αποφύγουμε οι μετανάστες να είναι θύματα δικτύων παράνομων διακινητών στην Ευρώπη. <clears throat> Η διαδικασία του Χαρτούμ είναι ένα στοιχείο, μια σφίδα σε μια συνολική στρατηγική. Κατανοώ τις ανησυχίες σας σε σχέση με τους στόχους αυτής της προσπάθειας. Παρ' όλα αυτά, θέλω να διευκρινίσω το ότι η πολιτική μας δεν αντιμετωπίζει τις, δεν θέλει να νομιμοποιήσει τις κυβερνήσεις της περιοχής ο στόχο μα είναι να θέσουμε τι κυβερνήσει αυτέ ενώπιον των ευθυνών του για να σωθούν ανθρώπινε ζωέ και να αντιμετωπιστούν οι διακίνητε. Πρέπει τα κράτη αυτά να τηρήσουν τι υποχρεώσει που έχουν αναλάβει. <clears throat> Είμαι σίγουρο ότι θα παρακολουθήσουμε και εσεί και εμεί τη διαδικασία από πολύ κοντά. Εξάλλου, το να ενισχύσουμε την ε, σύνδεση μεταξύ τη εσωτερική και τη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχουν συγκεκριμένε και συνολικές αντιμετωπίσεις για τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό είναι μια από τις προτεραιότητές μου. Θα αντιμετωπίσω τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Θεμετολόγιο της Μετανάστευσης που ανακοινώθηκε χθε μέσα στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2015. Επιπλέον. Καμία αμφιβολία δεν χωρεί ότι πρέπει να δώσουμε πιο ασφαλείς λύσεις για τα άτομα τα οποία έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Η Κομισιόν <clears throat> διερευνά αυτή τη στιγμή όλες τις δυνατότητες και ιδίως την δυνατότητα να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση για την ε, προσωρινή παροχή προξενικών θεωρήσεων ώστε να έρθουν οι πρόσφυγες στην Ευρώπη και να ζητήσουν άσυλο. Προς το παρόν, η ανα, ε, επανεγκατάσταση των προσφύγων είναι απαραίτητη μεταξύ μας. Αυτό πρέπει να είναι μια πράξη αλληλεγγύης που θα πρέπει να γίνει, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σώσουμε περισσότερες ζωές. Εφέτος ο αριθμός των θέσεων επανεγκατάστασης που έχουν δώσει τα κατημέλη έχει αυξηθεί. Ένα άλλο εργαλείο στη διάθεσή μα είναι τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και μέσα στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την υποστήριξή τη στις αφρικανικές χώρες, ώστε οι χώρες αυτές να μπορούν να υποδεχτούν μετανάστες στις καλύτερες, πρόσφυγες στις καλύτερες δυνατές Όπως είπα προηγουμένως, ούτως ή άλλως θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας και θα την παρακολουθήσουμε πολύ στενά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας, αλλά και για την παρουσίασή σας και τη δήλωση. Και τώρα ε, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον κύριο Ντέλα Παρακαλώ, Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους ε, ε, βουλευτές που πήραν το λόγο και που είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις εκτιμήσεις τους, τους προβληματισμούς τους και τις ανησυχίες τους όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας του Χαρτούμα. Εγώ θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο ανεφέρθη πανλημένος, δηλαδή το θέμα των στόχων και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διαδικασία του μου στόχο έχει να αναπτύξει μια τεχνική συνεργασία με τις αρχές ε, των χωρών της Ανατολικής Αφρικής και του κέρατος της Αφρικής. Όπως είπε ο Επίτροπος, βεβαίω δεν πρόκειται για νομιμοποίηση, δεν μπορεί να είναι από νομιμοποίηση των καθεστώτων αυτών των χωρών, αλλά ε, τεχνική συνεργασία που θα εστιάσει αυτή τη στιγμή σε δύο θέματα, στη διακίνηση ανθρώπων και στην διακίνηση μεταναστών. Ε, είναι αναμφίβολο ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσπαθήσουμε να σώσουμε τις ζωές μεταναστών που ξεκινούν επικίνδυνα ε, ταξίδια για να μπορέσουν να περάσουν ε, την Μεσόγειο, να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Ε, κυρίως θα πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτό το φοβερό έγκλημα της διακίνησης ανθρώπων, του δουλεμπορίου που γίνεται. αυτός είναι ο στόχος για την ανάπτυξη και για την εφαρμογή μιας τέτοιας συνεργασίας που μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς σε ευθυγράμμιση με άλλα θέματα της μετανάστευσης και της κινητικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι συνεπής στην βασική αρχή της πλήρου, του πλήρου σεβασμού των δικαιωμάτων των μεταναστών που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα μετανάστευσης. Θεωρώ ότι το να διευκολυνθούν οι επαφές με τις αρχές μιας σειράς χωρών με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν μέχρι στιγμής να ξεκινήσουν διάλογο, θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο για την ευαισθητοποίηση των εν λόγω χωρών για τα θέματα της προώθησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι ακόμα Κάτι ακόμα που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι η δήλωση αυτή επαναλαμβάνει την ανάγκη πλήρου σεβασμού των αρχών διεθνού προστασία. Πράγμα το οποίο τονίζει την σημασία να δοθεί προστασία στου πρόσφυγες και στου ετούντε άσυλο και βοήθεια στου μετανάστευς που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. Επίση, υπογραμμίζουμε την ανάγκη να αγγιηθούμε προστασία στου πρόσφυγε στου ετούντε άσυλο αλλά και στου εσωτερικά εκτοπισμένου Καθώ καθώς και να προσβλέψουμε και να τηρήσουμε τις αρχές τις διαδικασίες μάλλον ασύλου σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Άκουσα την έκφραση πολλών ανησυχιών και προβληματισμών τις οποίες δεν είμαστε ε, ε, αδιάφοροι, αλλά επαναλαμβάνω ότι το πρώτος μας στόχος είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Θεωρούμε πως είναι για μια ε, σοβαρή πρωτοβουλία που πρέπει να της δοθεί συνέχεια και θα πρέπει να γίνει. Βεβαίως θα πρέπει πλήρως να σεβαστούμε τις αρχές που ορίζονται στη δήλωση της Ρώμης ε, για την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας αλλά και για να αποφευθούν οι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν και τονίστηκαν. Πιστεύω πως είναι σημαντική η στήριξη από πλευρά των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η ενεργή συμμετοχή των κρατών μελών και επίσης πρέπει να υπογραμμίσω ότι τούτο εδώ το Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Και θα, σας διαβεβαιώ ότι θα ενημερώνεστε για τις εξελίξεις αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη δήλωσή σας, για την παρουσία σας και έχουμε έρθει